την ε, πρόταση της διάσκεψης των Προέδρων να υπάρχει η δημιουργία μιας ε, ειδική επιτροπής. Ε, η ψηφοφορία θα γίνει την Πέμπτη και όσοι έχουν να καταθέσουν τροπολογίες στη διάσκεψη των Προέδρων που θα γίνει η ψηφοφορία την Τετάρτη στις 7 η ώρα μπορούν να το κάνουν. Πάμε τώρα στο σχέδιο ημερίζες διάτραξης. Σύμφωνα με το άρθρο 809 οι ομάδες ζήτησαν η σημερινή συνεδρίαση να διαρκέσει μέχρι τις 10 η ώρα. Υπάρχουν αντιρρήσεις γι' αυτό? Οπότε γίνεται παράταση της σημερινής συνεδρίασης. Για την Τρίτη δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Πάμε λοιπόν στην Τετάρτη. Σύμφωνα. Παρακαλώ. Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω κάτι από την διάσκεψη των Προέδρων Μία από τις σημαντικότερες ευκαιρίες που έχουν οι βουλευτές είναι η δυνατότητα να εκφραστούν ε, στις παρεμβάσεις του ενός λεπτού για να εγείρουμε ζητήματα που σχετίζονται με την εκλογική μας περιφέρεια και αφορούν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν επαρκεί το ημίωρο που προβλέπεται για αυτή τη διαδικασία. Θα ήθελα να υποβάλω έτοιμα στη διάσκεψη των Προεδρών να παραταθεί στη μία ώρα παρακαλώ η διαδικασία των παρεμβάσεων του ενός λεπτού. Ευχαριστώ. Σήμερα στην ημερήσια διάταξη υπάρχει πρόβλεψη για ομιλία ενός λεπτού σχετικά με το θέμα. Μπορείτε μετά, σήμερα στην ημερήσια διάταξη έχουμε τις παρεμβάσεις ενός λεπτού. Μπορείτε τότε να μιλήσετε, υπάρχει πολλής χρόνος. Okay. Ωραία. Σε κάθε περίπτωση, ε, αν αλλάξει η μερίσια διάταξη θα το δούμε, αλλά σήμερα βλέπω ότι ε, δεν υπάρχει πρόβλημα και θα το συζητήσουμε και στη διάσκεψη των Προέδρων. Αλλά σήμερα με το ένα λεπτό που έχετε στη διάθεσή σας νομίζω ότι είναι αρκετό. Για την τρίτη λοιπόν δεν έχω κάποια πρόταση αλλαγής. Ε, τώρα για την Τετάρτη όσον αφορά στην ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία μετά από την βία του Ισλαμικού κράτους οι πράσινοι ζητούν μια αλλαγή του τίτλου και να, ο οποίος θα πρέπει να γίνει η ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και στη Συρία ειδικότερα μέσα στα πλαίσια του Ισλαμικού κράτους. Ο λόγος τώρα πηγαίνει στην, στον κύριο Άλιν Σμιθ. Ευχαριστώ. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι αμφιλεγόμενο αυτό. Θεωρούμε ότι είναι απολύτω δικαιολογημένο το ψήφισμα. Ε, το πιστεύουμε αυτό πρωτού το καταθέσαμε. Δείτε τη βία που ασκεί το ISIS. Ε, ε, φυσικά Βλέπουμε ότι υπάρχει μια τελείωτη σειρά θηριωδιών σε αυτές τις δύο χώρες ε, που έχουν επισύρει μια ανθρωπιστική κρίση ε, και πιστεύουμε ότι στο Ιράκ και στη Συρία θα πρέπει ε, κυρίως στο πλαίσιο του ίσης να αντιμετωπίσουμε τα ευρύτερα προβλήματα που υπάρχουν γιατί δεν υπάρχει μόνο το πρόβλημα της βίας του Ισλαμικού στρατού. Ελπίζω να αντιλαμβάνονται και να συμφωνούν οι συνάδελφοι με αυτή την αλλαγή. Που... Ευχαριστώ. Θέλει κάποιο να υπερψηφίσει, να καταψηφίσει ή να μιλήσει κατά αυτής της πρότασης, παρακαλώ. Δεν υπάρχει κάτι εναντίον. Ας ψηφίσουμε λοιπόν ποιοι υπερψηφίζουν. Ποιοι καταψηφίζουν. Αποχές εγκρίνεται. Για την Τετάρτη και το ΕΛΚ ζητά ε, να υπάρχει στη ε, στην διάταξη και ένα ψήφισμα για τους ε, διασυνδετητές ενέργειας. Η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ το λόγο στη θέση του συναδέλφου του κυρίου Μέλλου που δεν έχει φτάσει ακόμα. Θα ήθελε εδώ να προσθεθεί στη Σύνοδο Λομέλειας μία συζήτηση με ψήφισμα για τις διασυνδέσεις ενέργειας στα πλαίσια της περάτωσης της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Αγοράς. Το ευρωπαϊκό διαδίκτυο με τις διασυνδέσεις μου φαίνεται απολύτως αναγκαίο όχι μόνο για τις χώρες της Ιβηρικής Χερσονήσου αλλά και για τις χώρες της Βαλτικής. Είναι πολύ σημαντικό να λάβει γνώση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κατεπήγον τη ανάληψης μέτρων για αυτό το σκοπό. Ε, σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ελπίζω οι συνάδελφοι να στηρίξουν αυτή, αυτό το αίτημα. Ευχαριστούμε. Ποιο θέλει να πει κάτι πέρα αυτή τη ε, αίτηση, ο κύριο Μαρινέσκου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε καθορίσει πολύ σαφεί στόχου για τι διασυνδέσει τη ενέργεια. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νέα αγορά σε αυτόν τον κλάδο στην Ευρώπη και τα δίκτυα βρίσκονται ακριβώ στα θεμέλια αυτή τη νέας αγορά για να υπάρξει η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση. Γι' αυτό το ΕΛΚ υποστηρίζει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση για το θέμα. Ευχαριστούμε. Ποιο θα ήθελε να πει κάτι εναντίον αυτή τη πρόταση, ο κύριο Νίκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών διαφωνεί με το αίτημα αυτό με δύο πολύ για δύο πολύ λόγου. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει ήδη μια έκθεση πρωτοβουλία που καλύπτει αυτό το θέμα και θα υποβληθεί πολύ σύντομα. Και κατά δεύτερον, σε δύο εβδομάδες μόλις ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εύκοβιτ θα μας παρουσιάσει ένα ευρύτατο σχέδιο που καλύπτει αυτό τον προβληματισμό, το όλο θέμα των μεταφορών και των διασυνδέσεων. Κατά την άποψή μα το πρόγραμμα αυτό θα καλύψει ούτως ή άλλως το σύνολο του θέματος συμπεριλαμβανομένων των χωρών της Ιβηρικής Χερσονήσου και των χωρών της Βαλτική με ειδική μνήμα για τις χώρες της Μεσογείου και τα ανατολικά τη Ευρώπης. Νομίζω λοιπόν ότι καλό θα ήταν να περιμένουμε προηγουμένω το σχέδιο αυτό και να συζητήσουμε στην ε, Σύνοδο της 25ης Φεβρουαρίου το όλο θέμα. Είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα αυτό που θα μας υποβληθεί για του τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Αγοράς. Κύριε Λάμπερτ, θέλετε κι εσείς ε, να πείτε κάτι εναντίον. Παρακαλώ. Το είπατε πολύ νωρίς ε, και νόμιζα ότι θα ήσασταν υπέρ. Για να ψηφίσουμε λοιπόν. Ποιος είναι υπέρ της προτάσεως της κυρίας Γκροστέτ, παρακαλώ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Για την Τετάρτη έχω και μια σειρά από ε, συναδέλφους οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια πρόταση να προσταθεί στη δήλωση της Κομισιόν για την 70η επέτειο των ε, Συμφωνιών της Γιάλτας ένα ψήφισμα. Ο κύριος Μάρεκ Γιούρεκ έχει το λόγο για να ε, εμπεριστατώσει αυτό το αίτημα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσο βρισκόμαστε εδώ, Υπάρχει ε, η, επέτειος, η 70η επέτειος της διάσκεψης της Γιάλτα, όπου οι μισές χώρες της Ευρώπης είχαν την ελευθερία τους. Όμως ε, υπήρξε και μια ε, στρατιωτική απειλή για τις χώρες όπως η δική μου και χώρες της Βαλτικής που με στρατιωτικό τρόπο ε, τη στερήθηκαν και για τη Γερμανία ο, άνοιξε ο δρόμος για το διχασμό της, για τη διχοτόμησή της. Αυτό λοιπόν ε, το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να γίνει μια συζήτηση εις βάθος ε, για τις επιπτώσεις ε, στο παρόν της διάσκεψης της Γιάλτα. Και αυτό πρέπει να τελειώσει με ένα ψήφισμα. Ποιος θα ήθελε να πει κάτι υπέρ αυτής της πρότασης. Υπάρχει κάποιος που είναι εναντίον. Ο κύριος Λάμπερτς παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω όλοι συνειδητοποιούν τι σήμανε η διάσκεψη της Γιάλτας για την Ευρώπη, αλλά ας μην τα μπερδεύουμε όλα. Είμαστε εδώ πέρα σε ένα πολιτικό σώμα ερετών, δεν είμαστε ιστορικοί εδώ. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσουμε τα ιστορικά γεγονότα και να γράψουμε... Ε, ε, ιστορία, αλλά όχι για να εξυπηρετούμε τα συμφέροντα κάποιου. Να αφήσουμε την ιστορία στους ιστορικούς. Κάποιοι εδώ ενδιαφέρονται, αλλά νομίζω ότι δεν είναι πρόσφορο εδώ να κάνουμε συζητήσεις και ψηφίσματα για την ερμηνεία της ιστορίας. Δεν είναι η θέση μας αυτή. Ευχαριστούμε κύριε ε, Λάμπερτς, ο κύριος Ιστόφσκι. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλά και έχει συζητήσει ιστορικά γεγονότα. Την ε, εκατοστή επέτειο από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου τη συζητήσαμε επανειλημμένα και εφόσον προσυπογράφουμε όλοι τις αρχές ε, της ε, αλήθειας και της αλληλεγγύης δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε τη σημασία του διχασμού της Ευρώπης που επέσυρε η διάσκεψη της Γιάλτας και κατά 50 χρόνια είχαμε καθυστέρηση στην Ευρωπαϊκή Ενωπή. Αυτά είναι σημαντικά όχι μόνο για τη Βουλγαρία, τη Λετωνία, Λετωνία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Κροατία. Είναι κέρια σημασία σε αυτά τα ιστορικά γεγονότα για όλους ε, όσοι σέβονται ε, και ενστερνίζονται την αρχή της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Θα ήθελα να αποταθώ σε όλες τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου να απευθύνω μια διακομματική έκκληση. Ας μην επιδείξουμε αδιαφορία. Είναι ένα από τα πιο κέρια περιστατικά της ευρωπαϊκής ιστορίας. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε τη σημασία. Ας ψηφίσουμε λοιπόν ποιο είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήταν ξεκάθαρο ότι απορρίπτηκε. Ας το δούμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Έχουν ψηφίσει όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 82 υπέρ, 194 κατά, 30 αποχές, άρα απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην πέμπτη. Το ΕΛΚ ε, ζήτησε να ε, ολοκληρώσουμε την δήλωση της Επιτροπής ε, για την μάχη κατά της σεξουαλικής κακομεταχείρισης των παιδιών στο ίντερνετ με ένα ψήφισμα. Ο κύριος Χόλενμάιερ. Κυρία Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα προσπαθήσουμε άλλη μια φορά να ε, σας πω για ποιο λόγο το ΕΛΚ θέλει αυτό το πολύ δύσκολο θέμα της ε, σεξουαλικής ε, κακομεταχείρισης των παιδιών να επισφραγιστεί με ένα ψήφισμα. Μαζί λοιπόν με ένα κοινό ψήφισμα θα πρέπει μαζί με τη Συμμαχία των 50 χωρών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων ευρωπαϊκών χωρών ε, να ξεκαθαρίσουμε δημόσια ότι η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών θα πρέπει να είναι για μας ε, στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης παρά τα άλλα προβλήματα. Και μια κοινή στάση κατά αυτής της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών ε, αργότερα στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και με μια έκθεση πρωτοβουλίας και με άλλες πρωτοβουλίες ε, θα δείξει ότι ε, δεν καθόμαστε άπραγοι και παρακολουθούμε αυτά τα παιδιά που είναι θύματα κακοποίησης, αλλά εναντιονόμαστε σε αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε ένα κοινό χτύπημα, βαρύ χτύπημα σε αυτό το πρόβλημα. Κυρία Χολμάγερ, η κυρία Κοράτσα Μπίλτ θα ήθελε να μιλήσει για αυτό το αίτημα. Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει ούτε ένας γονέας ε, στην Ευρώπη που δεν ανησυχεί από τα νούμερα της Europol που μιλάνε από μόνα τους. Παιδιά κάτω της ηλικία των δύο ετών είναι θύματα βίας και κακοποίησης ή παρενόχλησης μέσω ίντερνετ. Αυτό που ζητώ κύριε ε, Πρόεδρε είναι να ε, υπάρχει ένα ψήφισμα διότι δεν μπορούμε να αρνηθούμε τις ανησυχίες των πολιτών της Ευρώπης. Δεν θέλω βέβαια από εξ αρχής να πω τι θα πούν οι συνάδελφοι κατά τη διάρκεια του ψηφίσματος. Υπερψηφίστε παρακαλώ, γιατί δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει κάποιος που θέλει να πει κάτι εναντίον αυτού του αιτήματο. Όχι. Για να ψηφίσουμε λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έτσι λοιπόν ε, το σχέδιο μερίσιας διάταξης ε, οριστικοποιείται. Ο κύριος Κλέτσος έχει το λόγο. Κλέζος έχει το λόγο. Αγαπητέ Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, προτείνω όπως ε, το σώμα μας απασχοληθεί ειδικά σε μια ειδική συζήτηση στην οποία θα προτείνετε εσείς και θα εγκρίνει το σώμα για την κατάσταση στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο αυτό ώστε να μην εκφράζει οποιοδήποτε απόψεις οι οποίες δεν εκφράζουν τις απόψεις του σώματος. Λυπούμε ιδιαίτερα διότι εσείς ο ίδιος αγαπητέ Πρόεδρε πήγατε στην Ελλάδα χωρίς να συζητηθεί το θέμα προηγούμενα στο σώμα. Τι εκφράζατε, απόψεις δικές σας, ατομικές ή απόψεις του σώματος ή απόψεις άλλων. Νομίζω ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη για την Ελλάδα και γι' αυτό είναι αναγκαίο και απαραίτητο να γίνει η συζήτηση. Θέλω να τονίσω, όπως έλεγα και προηγουμένως, ότι θα έρθει αυτή η μέρα όπου θα νικήσει ο ελληνικός λαός. Θέλω να τονίσω ότι όσοι προσπαθούν να εμποδίσουν τον ελληνικό λαό να αποκαταστήσει την εθνική του ανεξαρτησία και να την εμπεδώσει και όσοι θα προσπαθήσουν να τον εμποδίσουν να βγάλει τη θηλιά που του έχουν βάλει οι δανειστές θα σπάσουν τα μούτρα τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γκλέτσο. Η πρόταση για αυτή τη συζήτηση ήρθε λίγο αργά. Οπότε η ομάδα σας θα πρέπει να καταθέσει το αίτημα στη διάσκεψη των Προέδρων. Πηγαίνουμε λοιπόν τώρα στις ε, πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξάγεται στο πλαίσιο